So, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε αν θέλετε. Τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους σας αυτή την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Επιτροπή μας, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, σε ό,τι αφορά την ε, παρουσίαση των υποψηφίων για το βραβείο Ζαχάροφ από το 2018. Με το βραβείο αυτό τιμούμε τα άτομα τα οποία με τη δουλειά τους, με το έργο τους έχουν συμβάλει στην καταπολέμηση των αδικαιών και στην πρόσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλοι οι υποψηφοί έχουν ε, βάλει το στίγμα τους σε ό,τι αφορά το πλαίσιο αυτό στο διεθνή προσκήνιο. Θα ήθελα να σας επενθυμίσω ότι πρόκειται για την κίνηση, την αρχή της διαδικασία η επιλογή των υποψηφίων για το βραβείο Ζαχάροφ. 9 Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και θα υποβάλουμε μία λίστα, σύντομη λίστα τριών υποψηφίων στην διάσκεψη των Προέδρων και θα αποφασιστεί τελικά αυτό ε, στις 25 Οκτωβρίου. Το βραβείο Σαχάροφ είναι ενδεχομένω το πιο προβεβλημένο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τέτοιε βραβεύσει. Δεν είναι το μόνο ασφαλώ. Ε, λαμβάνουμε υπόψη διάφορε συνεργασίε που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα διάφορου μηχανισμού για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία πάντα θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο τέτοιων συμφωνιών με άλλε χώρε. Παρακολουθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στη σχέση με άλλες χώρες και κρίνουμε και τις αντιδράσεις των χωρών αυτών και θεωρούμε ότι μπορούμε να σημειώσουμε τη διαφορά, να έχουμε υπόψη ότι όποιος και να επιλεχθεί όλες αυτές οι περιοχές και οι χώρες αξίζουν την ε, προσοχή μας και την συγκεκριμένη δέσμευσή μας. Πρώτα δώσω το λόγο στον κύριο Παντσέρη για την υποτροπή ανθρώπινων δικαιώματων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιότητα ήταν 13 Σεπτεμβρίων και λάβαμε 8 άτομα ως υποψηφίους, 8 παρατακτές υποψηφιότητες. Θα βρείτε τα ονόματα στους φακέλους σας. Να δώσω το λόγο τώρα στον συνάδελφο τον κύριο Παντσερή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η παρουσίαση των 8 υποψηφίων είναι με αλφαβητική σειρά. Έχετε και ένα μικρό κείμενο για κάθε υποψήφιο και θα ήθελα να σας καλέσω όλους σας να παρουσιάσετε ο καθένας τον υποψηφίο του μέσα σε πέντε λεπτά. Κατά το όριο θα ακολουθήσει και μια σύντομη δελαγή απόψεων 10 λεπτά. Έχουμε χρόνο μέχρι τη μία και έχουμε διερμηνία μέχρι τη μία. Και προβλέπετε λοιπόν να ολοκληρώσω τη συνεδρία στη μία. Και να δώσω το λόγο στο Μάριο Μπουρκέτσι για την πρώτη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια μη κυβερνητική οργάνωση, την AfriForum, η οποία έχει ως σκοπό να προστατεύσει τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Νότια Αφρική με ιδιαίτερη επικέντρωση στα δικαιώματα των γεωργών. Η AfriForum λοιπόν προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε ό,τι αφορά τα θέματα δολοφονιών και εκτελέσεων των αγροτών και στα θέματα απολωτρίωσης της γης χωρίς αποζημίωση. Αυτή η πολιτική την οποία επιδιώκει η κυβέρνηση του ANC δεν ε, απειλεί μόνο τους ε, γεωργούς ε, αλλά και τους γεωκτήμονες ανεξαρτήτως εθνικότητας και αυτό ιδιαίτερα στα πλαίσια ενός ενδεμικού προβλήματος σε ό,τι αφορά το έγκλημα, ένα πολιτικό κλίμα ατιμορρησίας και ε, ενός κλίματος το οποίο προαγάγει τη βία κατά των αγροτών. Η Afri Φάρμα δημιουργήθηκε το 2006, είναι καταχωρισμένη ως μη κερδοσκοπική οργάνωση και σκοπό έχει την προστασία των δικαιωμάτων μιας μειονοτικής ομάδας. Αναγνωρίζεται διεθνώς για την προστασία των δικαιωμάτων της μειονότητας αυτής, προστατεύοντας ε, και τους αγρότες ως μια μεγάλη ομάδα του πληθυσμού της Νότιας Αφρικής. Υπάρχει και ένα μανιφέστο, ένας χάρτης ε, πολιτικών δικαιωμάτων για τις μειονότητες μπορείτε να το επισκεφτείτε online στο διαδίκτυο σε ό,τι αφορά διάφορα επίπεδα, σε επίπεδο οργανώσεων, κοινωνικό επίπεδο, πολιτικό επίπεδο, σε όλη την κοινωνία της Νότιας Αφρικής. του Αφριφόρουμ λοιπόν. Επικεντρώνονται ιδιαίτερα στους φόρους για την παραγωγή και όπου απειλούνται οι γεωργοί. Υπάρχει μια επίθεση λοιπόν κατά της ιδιωτικής εκμετάλλευσης και της, και της ιδιοκτησίας γεών. Και στην ε, Νότια Αφρική οι γεωργοί αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ζητήματα. Αυτό που είναι λοιπόν ξεχωριστό είναι ότι υπάρχουν πολιτικοί όπως ο γύρος Γιούλιος Μαλέμα, πρόεδρος του τρίτου μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος στην Νοτιοφρική, που ανοιχτά ε, πραγαγούν τη βία κατά των Γεωργών. Ο δεύτερος υποψήφιος είναι, ε, λέει ο πρόεδρος, είναι η κυρία Σίρνα Άτες, ε, η υποψήφια από την ομάδα του ECR, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους εκπρόσωπους της ε, ομάδος. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εκπρόσωπο των συναδελφων Hans Olaf Δεν είναι μόνο η ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών που έχουν υποβάλει την υποψηφιότητα τη κυρία Σέιραν Άντες. Είναι και άλλοι 40 ευρωβουλευτέ από διάφορα πολιτικά κόμματα. Η κυρία Σέιραν είναι δικηγόρο και ακτιβίστρια υπέρ των ανθρωπινών δικαιωμάτων γεννηθήσα στην Τουρκία. Μετέβησε η οικογένειά της στη Γερμανία όταν ήταν ακόμα παιδί. Καταπολεμά την ε, καταπίεση των γυναικών και αποτελεί σύμβολο κατά των ε, εκτελέσεων τιμής ε, κατά των γάμων παιδιών και άλλων πρακτικών που χαρακτηρίζουν το Ισλάμ έχει προφανώς προσελκύσει μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερα εχθρική ε, προσοχή. Έχει λάβει απειλές κατά της ζωής ε. της. Σε κάποια υπόθεση ο πελάτης της ε, δολοφονήθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά και η ίδια η κυρία Τέσος, δικηγόρος του ατόμου αυτού. Συνέχισε λοιπόν τη δράση της και έχει πραγματικά λάβει πολλές απειλές κατά τη ζωή της, ε, κατά τη ζωή της ίδιας της οικογένεια. Τον Ιούνιο πέρσι, με μεγάλο θάρρος ε, και τόλμη, ε, ήταν στα γένεια του Ινστιτούτ Γκέτε στο Βερολίνο συγγνώμη, ε, στα εγγένεια, ε, στην ε, παρουσίαση ενός τζαμιού, το οποίο αντίθετα με, το, με τα έθιμα του Ισλάμ μπορούν οι γυναίκες και οι άνδρες να προσεύχονται από κοινού. Το Τζαμί Ιμπν Ρουστ Γκέτε. Συναντήθηκα μαζί της τότε στο Βερολίνο και εγώ προσωπικά μπορώ να σας εγγυηθώ για την τόλμη και το θάρρος που χαρακτηρίζουν αυτή τη γυναίκα. Ξεκίνησε επίσης ε, την ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την κατάργηση του εξτρεμισμού και ένα σύμφωνο κατά του εξτρεμισμού στην Ευρώπη για να αντιμετωπιστούν τα πολιτικά παραθυράκια κατά του εξτρεμισμού για να υπάρχει ασφάλεια στην Ευρώπη. Έχουμε την αίσθηση λοιπόν ότι αν δεν το βραβείο Ζαχάροφ θα ήταν μια πολύ αρμόζουσα κίνηση σε ό,τι αφορά την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία, την ανεξιθρησκεία, τα οποία εκπροσωπεί. Γι' αυτό και υποστηρίζω την εξαιρετική αυτή υποψήφια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, ο επόμενος υποψήφιος είναι ο Σέζαρ της ομάδας Άλντε των Φιλελευθέρων. Η κυρία Σάκε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να παρακαλέσω να μου χαρίσετε την προσοχή σας για να σας μιλήσω για τον κωδικό Σίζαρ. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε την ε, πραγματική ταυτότητα του προσώπου αυτού και θα κατανοήσετε γιατί σε λίγο. Ο Σίζαρ Κέσσαρ δηλαδή ε, υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας ε, των βαρύτατων ε, εγκληματικών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Συρία και μπόρεσε να τα ε, φωτογραφίσει με πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο για τον εαυτό του και την οικογένειά του μπόρεσε να εξαγάγει λαθρέα 55.000 φωτογραφίες που έχουν καταγράψει βασανιστήρια και, και θάνατο 11.000 σύρων έγινε και έκθεση εδώ στο Κοινοβούλιο όπου δείξαμε τις φωτογραφίες αυτές και οι φωτογραφίες αυτές μιλούν από μόνες τους. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές ό,τι αφορά την βαρβαρότητα και τις βαρβαρότητες που έχουν γίνει στην Συρία. Η Human Rights Watch έχει ε, επαληθεύσει την εγκυρότητα των φωτογραφιών αυτών, το οποίο λέει πολλά. Το ΔΕ Μουσείο του Ολοκαυτώματος στι Ηνωμένε Πολιτείε έχει εκθέσει τις φωτογραφίες που μπόρεσε να εξαγάγει λαθρέα ο Κέσαρ από την Συρία. Είμαι πεπισμένη ότι κάποια μέρα όπου οι Σύροι θα αποδώσουν ευθύνε, οι φωτογραφίες του Σέζαρ θα αποτελέσουν ε, σημαντικό μέρος ε, των ε, πιστηρίων. Είμαι βέβαια ότι ο Σέζαρ είναι πραγματικός ήρωας, ένας απλός σύρος, καθημερινός σύρος, ο οποίος έλαβε μια θαραλέα απόφαση ε, ε, εν ώψη βαρύτατων παραβιάσεων ε, των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τις στρατιωτικές συριακές δυνάμεις και βέβαια από το κράτος. Και χέρι εκτιμήσεως από όλους τους σύρους για, το, για αυτό που έχει κάνει. Χθες η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο στο όνομά του και θα είναι ορθό, θεωρώ, εμείς ως Ευρωπαίοι να αναγνωρίσουμε τις ηρωικές πράξεις του ε, Σέζαρ και να αναγνωρίσουμε επίσης ότι ακόμη διατρέχει σοβαρότατο κίνδυνο διότι το καθεστώς Άσαντ εξακολουθεί να διώκει τους αντιπάλους του ακόμη και ολόκληρες δεκαετίες μετά από τις πράξεις τους. Έχουμε ένα σύντομο τώρα βίντεο για να μπορέσετε να ακούσετε τα λόγια του ίδιου του Σίζαρ και ε, με τον τρόπο αυτό λύγει και η παρουσίαση της υποψηφιότητάς του. Κάθε άνθρωπος έχει ένα απόθεμα υπομονής και για τρία χρόνια φωτογραφίζουμε τα σώματα των αθώων που σκοτώνονται κάθε μέρα. Και ήμουνα τόσο φοβισμένος κάθε πρωί που χαιρετούσα τη γυναίκα μου. Φανταζόμουν ότι μπορεί να μην την ξαναδώ. Οπότε ναι, με επηρέασε. Γιατί έβλεπα παντού πάρα πολύ οδύνη. Αλλά είτε εγώ είτε οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος που έβαλε τη ζωή του σε κίνδυνο και έθεσε και την ζωή του της οικογένειας και των φίλων και των παιδιών του σε κίνδυνο, αλλά ξέρει στην καρδιά του πως αν έχει, αν έχει έστω και μια σταγόνα ε, ανθρωπισμού στην καρδιά του, δεν μπορεί να γυρίσει το πρόσωπο και να μην παρουσιάσει τι γίνεται. Οπότε τι το έκανε. Όταν τελειώναμε τη δουλειά, τελειώναμε το βράδυ, έπαιρνα όλε τι φωτογραφίε και όλα τα αρχεία από τον υπολογιστή του γραφείου της στρατιωτικής αστυνομίας και τα βάζα σε πολύ μικρά στικάκια, πολύ μικρά σε μέγεθος και σε κάρτες μνήμης. Και μετά πήγαινα σε άλλο σημείο μακριά από το ε, γραφείο και είχα ένα φίλο εκεί ο οποίος έπαιρνε αυτά τα στικάκια, τα φόρτωνε στον προσωπικό του ε, υπολογιστή και με τον τρόπο αυτό καταφέρναμε να ξεφύγουμε κάθε μέρα. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί περνούσα συνέχεια από σημεία ελέγχου, checkpoint όλη την ημέρα. Ε, ήταν τα στρατιωτικά, καθεστωτικά αυτά σημεία και μου έκαναν πάρα πολλούς ελέγχους. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Ο τέταρτος υποψήφιος είναι ο Γιάνν Τζόνσον. Και εδώ θα δώσω το λόγο καταρχήν στον κύριο Καστάλδο για να μας τα παρουσιάσει. Να σας πω πως μέχρι την τελευταία μου πνοή θα δώσω τη μάχη. Ο Ντουέιν Τζόνσον το φώναξε αυτό και είναι πολύ ηρωική αυτή η ε, δήλωσή του σε αυτό το σχολείο του Αγίου ε, Φραγκίσκου και για τον οποίο ε, ξέρουμε ότι πήγε τη Μονσάντο στα δικαστήρια. για το πολύ αυτό τοξικό ε, που θα μπορούσε να τον είχε σκοτώσει και που έβαζε σε κίνδυνο την ζωή των παιδιών στο σχολείο που δούλαβε. Και είχε αυτά, ε, αυτές τις κοιλίδες στα χέρια του όταν χρησιμοποίησε το ζυζανιοκτόνο που έδειχνε ότι υπάρχει κάποιο βασικό πρόβλημα που ήταν καρκίνος αιματολογικός που προκλήθηκε από την επαφή. Και συνέχεια του κάναν τηλεφώνα με υποσχέσεις από τη Μονσάντο, αλλά ποτέ αυτές οι υποσχέσεις δεν ε, ε, δεν ε, έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Και όταν του είπε κάποια μέρα ο εργοδότης ότι κοίταξε να δεις, δεν θα κάνουμε τίποτα, πήγε στα δικαστήρια και έδωσε τη μάχη με το χαμόγελο, ακόμα και όταν νόμιζε πως όλα είχαν χαθεί. Αυτός ο γίγαντας της αγροχημικής βιομηχανίας κατάφερε να παρακάμψει την επιστημονική κοινότητα και κάποιες επιστημονικές εκθέσεις για το ζυζανιοκτόν αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι αντίστοιχο με το ότι κάνανε η βιομηχανία του καπνού τη δεκαετία του 50 για να μην γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα του καπνίσματος και αυτός συνέχισε παρόλο που λόγω χημειοθεραπείας ήταν πολύ αδύναμος και η γυναίκα του χρειάστηκε να δουλεύει 14 ώρες την ημέρα σε δύο δουλειές για να μπορεί να πληρώσει για όλα σε αυτούς τους γιατρούς. Υπέφερε, πόναγε και νομίζω ότι θα πρέπει να τιμήσουμε το θάρρος του 280 εκατομμύρια δολάρια χρειάστηκε να πληρώσει Μονσάντο, ιστορική απόφαση δικαιοσύνη και είναι πραγματικά παράδειγμα για θύματα τα οποία κινδυνεύσαν και έχασαν την υγεία τους γιατί κάποιοι έβαλαν το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη υγεία. Είναι μια θαραλέα φωνή και νομίζω ότι αξίζει ε, το βραβείο Ζαχάροφ για το 2018. Ο Ντουέιν Τζόνσον δεν είναι μόνο ένας κυπουρός από την Αμερική με τρία παιδιά αλλά ένας από τους εκατοντάδες ασθενείς ε, με καρκίνο που κατήγγυλαν τη Μονσάντο γιατί ε, έβαλε το κέρδος της πάνω από την υγεία τους. Ήταν, κόντεψε να, πεθάνει, έχει λέμφωμα και δεν μπορεί να δουλέψει. Και αυτό έγινε γιατί χρησιμοποίησε το Roundup, αυτό το προϊόν ε, με γλυφοσάτη τη Μονσάντο, κατά την κυπουρική του εργασία. Και τους πήγε στο δικαστήριο γιατί πιστεύει ότι η ουσία αυτή προκαλεί καρκίνο. Και καταδικάστηκε η Μονσάντο σε μια τεράστια αποζημίωση 270 εκατομμύρια δολάρια ύψωσε το ανάστημά του εκφράζοντας τους χιλιάδες που έχουν ασθενήσει και είπε ο δικαστής ότι είναι κακοήθηση η πράξη της Μονσάντο χρόνια προσπαθούν να πείσουν τους χρήστες και τους πολιτικούς πως υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία και αποδεικνύουν πως το Roundup και η γλυβοσάτη όντως προκαλούν, προξενούν καρκίνο. Δεκαετίες κερδών για μια πολυεθνική, αλλά χάρη στον Dwayne Johnson πια δεν γελάει η Μονσάντο, γιατί τους προτείνουμε. Προτείνουμε τον άνθρωπο αυτό για το βραβείο Ζαχάροφ, γιατί δεν θέλουμε μόνο να τιμήσουμε ε, τον άρρωστο Δαβίδ κατά του ε, μεγάλου ε, Γολιάθ, αλλά γιατί θέλουμε ε, να τιμήσουμε όσους μάχονται τις, τις πολυεθνικές και υπάρχει το εξής. Δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος που πεθαίνει από καρκίνο, αλλά είναι ένας άνθρωπος που αποδεικνύει τι σημαίνει γλυφοσάτη που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες σε όλο τον κόσμο. Και περνάει η ουσία αυτή στο έδαφος, στον αέρα, στα ύδατα. Είδατε τι έκαναν οι αρχές της Ε, βρήκαν υπολείμματα ακόμα και στη βροχή. Είναι παντού και είναι αναπόφευκτη. Η αναγνώριση λοιπόν του κινδύνου και η ανάληψη ευθύνης είναι απαραίτητες για χιλιάδες κόσμου και το να τιμήσουμε τον άνθρωπο αυτό θα ξεπερνούσε την απλή υποψηφιότητα ενός μεμονωμένου ανθρώπου και θα έδινε θάρρος σε όσους έχουν υποστεί αυτές τις τεράστιες επιθέσεις από τις πολυεθνικές, θα τους προσέφερε ε, ελπίδα για το μέλλον. Το 11 ONG Να σας πω πως ε, έχουμε και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έχουν, ε, κάνουν διάσωση στη Μεσόγειο, είναι υποψηφιότητα από τους σοσιαλιστές και έχουμε εδώ ε, τους ευρωβουλευτές που θα μιλήσουν γι' αυτό. Οι σοσιαλιστές έχει την τιμή να παρουσιάσει την υποψηφιότητα των ε, που σώζουν ζωές στη Μεσόγειο. Είναι μια υποψηφιότητα συλλογική με 11 ΜΚΟ, οι οποίες πραγματικά πήδηξαν στη θάλασσα κυριολεκτικά από το 2015 για να σώσουν ανθρώπινες ζωές και για να καλύψουμε ένα τεράστιο κενό που άφησαν οι κυβερνήσεις και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Είναι το πιο ανθρώπινο πρόσωπο της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι ένα συγκεκριμένο χέρι βοήθειας που προσφέρει βοήθεια εκεί που χρειάζεται το διεθνέ δίκαιο, τα διεθνή δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία βεβαίω είναι στοιχείο κλειδί για να του ντυθεί το Ζαχάροφ. Και έχουν ε, απαγγελθεί κατηγορίε κα... κα... κατηγορίες δικαστικές, έχουν διωχθεί και καμία, κανένα ε, σκάφος δεν πλέει σήμερα στην Κεντρική Μεσόγειο γιατί δεν τους επιτρέπουν παρόλο που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη αυτή η θάλασσα. Θα πρέπει η ευρωπαϊκή κοινωνία να στηρίξει όσους εξ ονόματος τους μας βοηθάνε να ε, υποστηρίξουμε τις αρχές μας και τις αξίες μας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να δώσουμε το ζαχάρο σε αυτές τις ΜΚΟ θα είναι σαν να μιλάμε για τους εαυτούς μας, σαν να είμαστε εμείς το στόχο και να αναγνωρίσουμε πως κάναμε λάθος και να δημιουργήσουμε πίστη και πεποίθηση στην αλληλέγγυη Ευρώπη που όλοι στηρίζουμε. Όποιο θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο για να υπερασπιστεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα πρέπει να στηριχθεί και όχι να διώκεται. Αυτή είναι η Ευρώπη στην οποία πιστεύω, είναι η Ευρώπη στην οποία πιστεύουν η πλειοψηφία των πολιτών μα. Για αυτήν την Ευρώπη θέλουμε να δώσουμε τη μάχη και γι' αυτό σα ζητώ να στηρίξετε αυτή την υποψηφιότητα για το βραβείο Ζαχάροφ του 2018, η ΜΚΟ που σώζουν ζωέ στη Μεσόγειο. Estoy muy honrada de presentar al Premio 2010. Χαίρομαι που μπορώ να παρουσιάσω και από τους πράσινους αυτή την υποψηφιότητα. Οι Open Arms και άλλοι, 11 συνολικά, που σώζουν ζωές μεταναστών στη Μεσόγειο. Όταν ανέβηκα στο σκάφος, Open Arms απέναντι από τις λιβικές αρχές, είδα πρώτο χέρι πόσο ηρωικές προσπάθειες κάνει το πλήρωμα. Είδα πώς οι διασώστες, οι ε, γιατροί, οι νοσοκόμες, οι εθελοντές, όλοι έπεφταν στον, στο νερό για να σώσουν ζωές. Σώζαν την τιμή της Ευρώπης, γιατί είναι ντροπή ε, να αφήνουμε να πνίγεται ο κόσμος. Θα σας δείξω αυτό. Ξέρετε τι είναι, πιστεύετε πως αυτό μπορεί να σώσει ζωής. Ξέρετε τι γράφει πάνω, πως δεν σώζονται ζωές, μην αφήνετε να φοράνε ε, αυτό τα παιδιά όταν μπαίνουν στη θάλασσα. Και αυτό βρέθηκε σε μία βρέθηκε σε μια παραλία της Λέσβου και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι όταν βρίσκεις ένα οποιοδήποτε τέτοιο γυλαίκο ε, κάπου στη θάλασσα έχει πνιγεί ένα παιδί. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ε, σώζουν όχι μόνο ζωές αλλά την αλληλεγγύη της αξίας μας και όλες οι οργανώσεις που ε, είναι οι υποψήφιες σήμερα έχουν ποινικοποιηθεί, έχουν διωχθεί, τους έχουν πάρει τα σκάφη, τους έχουν κλείσει στα λιμάνια και αυτή τη στιγμή το μόνο ε, σκάφος, το Aquarius που κάνει διάσωση είναι υποδίωξη σε ένα από τα κράτη-μέλη. Και ξέρουμε πως υπάρχουν πολύ καλές υποψηφιότητες και πολλές εκτός Ευρώπης. Αλλά για μια φορά θέλουμε κι εμείς να πάει αυτό σε μια μη κυβερνητική οργάνωση Ευρωπαία, γιατί θα πρέπει εμεί να διασώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη, που πλήττονται από αυτή την τραγωδία, να είμαστε άνθρωποι και να δώσουμε μια ευρωπαϊκή απόκριση. Ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη και ας έχουμε το θάρρος και την ευθυξία να είμαστε ακόμα άνθρωποι. Και ίσως το βραβείο αυτό θα βοηθήσει να σώσουμε ζωής, γιατί αυτό το γυλαίκο δεν θα σώσει ζωές, αλλά αυτά τα σκάφη σώσουν ζωές και θα μπορέσουν έτσι να συνεχίσουν τη δουλειά που κάνουν. Ε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφε και ας περάσουμε τώρα στον έκτο υποψήφιο Όλεξ Σέντσοφ υποψηφιότητα που καταθέτει η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με υπερηφάνεια παρουσιάζω εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τον υποψήφιό μας για το βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το, που φέρει το όνομα του επιστήμονου Ζαχάροφ. Είναι ο κύριος Σέντσοφ. Θεωρούμε ότι η, ειρηνική του διαμαρτυρία κατά της ρωσικής κατοχής στην Κρυμαία και ο αγώνας για την απόλυση των Ουκρανών πολιτικών κρατουμένων αποτελούν ε, αγώνα υπέρ της ελευθερίας σκέψεως. Ο Όλεξ γεννήθηκε το 1976. Είναι Ουκρανός ε, σκηνοθέτης που ε, γεννήθηκε στην Κρυμαία και εκτεί ποινή 20 χρόνων κάθεξης σε ρωσική φυλακή. Είναι ο γνωστός για διάφορα ντοκιμαντέρ που έχει γυρίσει και ιδίως από το 2011 συνελήφθη το 2014 επειδή αντιτάχθηκε στην ε, ρωσική προσάρτηση της Κρυμαίας. Το 2015 καταδικάστηκε από ρωσικό δικαστήριο σε 20 χρόνια κάθερξη. Η απόφαση αυτή, η καταδίκη δηλαδή αυτή, χαρακτηρίστηκε άδικη και στηριγμένη σε ψεύτικα στοιχεία. Ο Όλεξ Σέντσοφ είναι αθώος βρίσκεται στη φυλακή παραπάνω από τέσσερα χρόνια. Από τον Μάιο φέτος κάνει ε, απεργία πείνας. Ζητεί από τις ρωσικές αρχές να απολύσουν 70 ε, Ουκρανούς κρατουμένους στη Ρωσία ή στην Κρυμαία για λόγους πολιτικούς μετά από την προσάρτηση της Κρυμαίας. Δεν ζητεί καν τη δική του απόλυση. Ο Λεξέντσοφ αποφάσισε να απευθύνει αυτή την έκκληση με την ελπίδα ότι θα ακουστεί η φωνή του και ότι θα ισχύσουν οι αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Πιστεύει στην υπεροχή του δικαίου απέναντι στην ομή και στην εξαπάτηση και αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για κρατούμενο συνείδησης. Έχουν περάσει πάνω από 100 ημέρες απεργίας πείνας. Η υγεία του είναι σε μεγάλο κίνδυνο με την στήριξη στον Όλεγ Σέντσοφ εμένουμε και επιμένουμε στις πεπιθήσεις μας για τις παγκόσμιες ισχύω αρχές της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της ελευθερίας σκέψης. Αυτή η ελευθερία σκέψης είναι και ο μεγάλος εφιάλτης όλων των δικτατόρων και αυταρχικών καθεστώτων που δεν τους επιτρέπει να ελέγξουν τον κόσμο και Επομένω, είναι και το καλύτερο όπλο για να αντιμετωπίσει κανεί του δικτάτορε αυτέ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την ελευθερία να πεθάνει σε σιγή. Θα είναι ο κύριος Σέντσοφ ο πρώτος που θα τιμηθεί με βραβείο Ζαχάροφ από την Κρυμαία, προχώμενος από την Κρυμαία. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση της υποψηφιότητας. Ο έβδομος υποψήφιος είναι η Μέρι Βάγνερ, την οποία, η υποψηφιότητα της οποίας προτείνουν ο Μάρεκ Γιούρεκ και 41 άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δίνω το λόγο στον κύριο Γιούρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος ε, διαφόρων μελών πολιτικών ομάδων αλλά και ανεξαρτήτων βουλευτών έχω την τιμή να ε, προτείνω την υποψηφιότητα της Μέρι Βάγνερ που είναι Καναδί και ε, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των αγενήτων. Οι διαμαρτυρίες οι οποίες έχει προβεί είναι πάντοτε απολύτως ειρηνικές. Δεν έχει επιτεθεί εναντίον κανενός. Άλλοι επιτίθεται εναντίον της και μάλιστα έχει, ε, την έχουν βάλει και στη φυλακή. και ε, φέρει ε, η ίδια στους ώμους της τον σταυρό της ε, άδικης δικαιοσύνης. Στηρίζει τους πιο αδύναμους και στηρίζει και το δικαίωμα έκφρασης. Άλλωστε, ε, η αξίζει, αξίζει να υποστηριχθεί η υποψηφιότητά της από όλους και από αυτούς που έχουν συνυπογράψει ε, τις διακηρύξεις του ε, Ρομπέρ Σουμάν, του Αλτσίδε Τιγκάσπερη, που είναι και το τιμόμενο πρόσωπο στην αίθουσα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ να ακούσετε την ε, μαρτυρία της ίδιας της Μέρι Βάγνερ. from across Χαιρετισμού έχετε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ονομάζομαι Μαρι Βάγκνερ και μου ζητήθηκε να σα πω δύο κουβέντε. Είμαι Καναδί με Ιρλανδικέ ρίζε από την ε, πλευρά τη μητέρα μου. Από τότε που θυμάμαι, προσπαθούσα να αποτελέσω τη φωνή για του ε, μικρού αδερφού και, ε, και αδερφέ μα που διακινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή του μέσα στη μητέρα τη μητέρα του. Από, την... από τότε που ήμουν 20 χρονών και ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια. Έχω περάσει πέντε χρόνια στην φυλακή για λόγω τη ειρηνικής μου δράση, εξ ονόματο των αγέντων αυτών παιδιών και των μητέρων του, που ε, καθημερινά φροντώνονται. Επανελειμμένα με έχουν κατηγορήσει για απάτη, για την παρεμπόδιση ε, άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων και επίσης ε, επειδή δεν απάντησα στις, ε, δεν ε, ανταποκρίθηκα στις ε, εντολές να μείνω μακριά από τέτοιες κλινικές. Η Λίντα και εγώ έχουμε ξεκινήσει λοιπόν το, τη διαδρομή αυτή, όχι μόνο επειδή πιστεύουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά επειδή πιστεύουμε και στα λόγια του Ιησού, που είπε ότι κάνει στους αδερφούς μου το πράττεις και σε μένα, ότι δεν δίνεις στους αδερφούς σου, δεν δίνεις και σε μένα. Από την εμπειρία μου, έχοντας συνομιλήσει με εκατοντάδες γυναίκες ε, που υποφέρουν λόγω των ε, αμβλώσεων που έχουν υποστεί, τίποτα δεν μπορεί να απέχει πιο πολύ από την αλήθεια. Η, η άμβλωση ε, τραυματίζει βαθιά τη γυναίκα. Όταν ναι, μια γυναίκα κάνει μια έμπλωση συνενεί στην δολοφονία του παιδιού τη και σε κάποιε περιπτώσει εξαναγκάζεται να το κάνει αυτό. Δεν είναι δικαίωμα, είναι μια απόλυτη ήττα για τη γυναίκα, γιατί είναι η μητέρα ενό μικρού παιδιού. Έχει δοθεί ένα μήνυμα ότι το μωρό τη δεν αξίζει να το υπερασπιστεί. Και έτσι λοιπόν πρόκειται για μια επίθεση κατά της μητρότητας, ε, της πουλάνε ένα ψέμα το οποίο δεν πρέπει να επιλύσει το πρόβλημά της, γιατί το πρόβλημα δεν είναι το μωρό, το πρόβλημα είναι οι συνθήκες οι οποίες είναι εκδικές στην υποδοχή αυτής της νέας ζωής. Ε, κάθε μία τέτοια λοιπόν, ε, τέτοια, μια, κάποια νέα τέτοια ζωή ε, καλεί στον κόσμο να δημιουργηθεί θέση για αυτήν και η απάντηση θα πρέπει να είναι αγάπη και βοήθεια όχι η βέη καταστροφή της ζωής. Μόλις λοιπόν απαρνηθούμε αυτή την αρχή ότι κάθε ανθρώπινη ζωή είναι ιερή, ποιανού η ζωή μπορούμε να αγγιηθούμε γιατί είναι η πιο ευάλωτη αυτή η πολίτες η οποία είναι υποκίνδυνο και βέβαια κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ασφαλής πλέον ο πρόεδρος. Σχόλια παρακαλώ δεν υπάρχει περιθώριο για σχόλια, μάλλον α, δεν α, απαγορεύονται τα σχόλια, αυτή είναι προφανή. Και θα δώσουμε τώρα το λόγο του υπευθύνους της ΓΚΟΕ για τον τελευταίο υποψήφιο, τον κύριο Νάσερ Σεφτσάβη. Υποψήφιο υποψήφιος, όπως σας είπα, από την ΓΚΟΕ και 39 άλλων μελών. Η κυρία θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το Μαρόκο είναι μια μεγάλη και όμορφη χώρα με πλούσια ιστορία σε ό,τι αφορά όμως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η συμφωνία του 1799 ήταν αυτή που μας έδωσε μεγάλη ελπίδα και η καθυστερημένη υλοποίησή της επίσης. Αλλά δυστυχώς αυτά δεν δεν μεταφράζονται στην πράξη και κυρίως όχι σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, όπως αποφανθήκε και η σχετική επιτροπή του Μαροκινού Κοινοβουλίου. Οι ανισότητες κοινωνικές, η ανεργία των νέων, η φτώχεια εξηγούν αυτή την αύξηση της δημόσιας κατακραυγής. Ωστόσο, το θέμα του Ιράκ, το κίνημα του Ρίφα, ε, το οποίο τον Οκτώβριο του 2016 έχει καταγγείλει αυτά τα περιστατικά. Και έτσι σε πολλές περιστάσεις ε, αποκρισταλώθηκε αυτή η δημόσια καταγραφή. Υπάρχει μεγάλη ιστορία λοιπόν ε, αντίστασης υπό την κατοχή της Γαλλίας, της Ισπανίας τη δεκαετία του 50 και θεωρούμε ότι ε, έχει εγκαταλειφθεί ο λαός του Μαρόκου από τις κεντρικές εξουσίες ε, και στην Ήπεθρο το 85% του κόσμου δεν έχουν καν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Και έχουμε λοιπόν μια τέτοια πλούσια παράδοση για την... Ε, μετά το θάνατο του και οι οι ειρηνικές διαδηλώσεις, άνθρωποι με ένα λουλούδι, με ένα κερί πολλαπλασιάστηκαν και οι μαροκινές ε, αρχές ανταποκρίθηκαν με μέτρα καταπίεσης. Και Ξεκίνησαν δικαστικές διώξεις κατά όλων και κατά των δημοσιογράφων που ήθελαν να καλύψουν τη διαδικασία και τα περιστατικά αυτά ακόμα και ανηλίκων οι οποίοι κατηγορήθηκαν για σεπερατισμό, για τρομοκρατία παρόλο που το μόνο που ζητούσαν ήταν να υπάρχουν πανεπιστήμια, να υπάρχουν νοσοκομεία και κοινωνική δικαιοσύνη και έχουν δημοσιευτεί πολλές ε, σχετικές παγκόσμιες μελέτες για την κατάσταση στις ε, φυλακές παρά το γεγονός ότι το Μαρόκο έχει προσυπογράψει την Εθνή Συνθήκη κατά των ε, βασανιστήριων και ο Νασέρ Ζευζάφ ήταν από τους ακτιβιστές του Ιράκ τον παρουσιάζουμε λοιπόν την υποψηφία του σήμερα. Και μετά την τηλεφωνία του ψαρά Μοξίν Φίκρη εξέφρασε την αντίθεσή του και στις 29 Μαΐου του 2017 ε, συνελήφθησε, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση και Πέρασε από πολλά βασανιστήρια. Υποστηρίζοντα λοιπόν την υποψηφιότητά του, δίνουμε ένα μήνυμα προς τις μαροκινές ε, αρχές. Ένα μήνυμα ότι η καταστολή δεν θα βοηθήσει. Αντιθέτως, ε, και πολλά έχουμε ακούσει τους τελευταίους μήνες, ε, έχει καταφτάσει στην Ισπανία και ζήτησε άσυλο στην Ισπανία. Υπάρχουν λοιπόν αυτέ ε, τα κατηγορώ κατά των μαροκινών αρχών που καταπιέζουν την μαροκινή νεολαία. Ναι, Θα πρέπει να βοηθήσουμε το Μαρόκο για να ανταποκριθεί στις ε, ανάγκες του λαού της και να ανανεώσει τους δεσμούς με το παρελθόν τους. Δεν υπάρχει δικαιολογία να υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι και βασανιστήρια στο σημερινό Μαρόκο και γι' αυτό λοιπόν σας καλώ να ψηφίσετε υπέρ της συμβολικής αυτής υποψηφιότητας του να σε ζευσαφή. Σας ευχαριστούμε Μαρή Κριστίν, λέει ο Πρόεδρος. Και έτσι ολοκληρώσαμε την παρουσίαση των υποψηφίων για το βραβείο Ζαχάροφ. Έχουμε λίγο χρόνο για ομιλία. Ένα λεπτό κατά το όριο όμως. Η κάτι πυρηνή πρώτη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω πως στηρίζω τον Νάζερ Σαφσάφιος, πραγματικά εξαιρετικό άνθρωπο που στην, στο κίνημα του Ρίφ στο Μαρόκο ε, ύψωσε τη φωνή του με ειρηνικό τρόπο μέσω του κινήματός τους για παιδεία, για υγεία, για περίθελψη και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει πολύ έντονη πίεση από τις μαροκινές αρχές του ΡΙΦ. 41 ανήλικοι, 800 συνολικά ε, άνθρωποι μπήκαν φυλακή ε, και κάποιοι καταδικάστηκαν από το ΧΙΡΑΠ και στα περίπου 20 χρόνια ε, και πρέπει να σας πω είναι ένα μήνυμα και για το Μαρόκο και για τη διασπορά του Μαρόκου που ζει στην Ευρώπη αλλά και για τη μαροκινή κυβέρνηση πως δεν τους ξεχνάμε και θα συνεχίσουμε τη μάχη μας κατά της αδικίας μέχρι να έχει απελευθερωθεί και ο τελευταίος πολιτικός κρατούμενος. Και τέλος, επιτρέψτε μου, θα ήθελα να τιμήσω τους γονείς ε, του ανθρώπου αυτού που ήρθαν από το Μαρόκο στις Βρυξέλλες σήμερα και κάθονται εκεί πίσω και να τους ευχαριστήσω όχι μόνο την ΚΟΕ, αλλά και τα 43, τους 43 ευρωβουλευτές που υπέγραψαν την υποψηφιότητα αυτή. Ευχαριστώ, κύριο Μιράντα. Κυρία Μιράντα, με συγχωρείτε, ευχαριστώ πολύ. Υπενθυμίζουμε πως η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πως η άμβλωση είναι απόλυτα, ε, απόλυτο δικαίωμα των γυναικών και γι' αυτό καταδικάζουμε με περηφάνεια, γιατί πραγματικά ήταν απέσιο να ακούς κάποια πράγματα εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο, το γεγονός πως το δικαίωμά μας αυτό το ουσιαστικό πλήττεται. Έχουμε αυτό το δικαίωμα της επιλογής. Και λυπόμαστε πάρα πολύ αυτή την υποψηφιότητα της Mary Wagner, γιατί θεωρούμε πως είναι μια χειραγώγηση του βραβείου για ε, εξτρεμαστικούς ε, ιδεολογικούς σκοπούς και που δεν τιμά και τους προηγούμενους που έχουν βραβευτεί. Ευχαριστώ πολύ να τονίσω κι εγώ. Είναι η κυρία Ατές η δική μας υποψηφιότητα. Είναι υπέρ της ελευθερίας του λόγου που ακολουθεί μια διαφορετική ε, προσέγγιση προς το Ισλάμ. Θα ήθελα να μιλήσω στο στόχο για τον οποίο δίδεται το βραβείο Ζαχάροφ και ξέρω πως έχουν περάσει διάφορες αλλαγές τα τελευταία χρόνια, αλλά η πρώτη προτεραιότητα, η αρχική προτεραιότητα και ο πρώτος στόχος σήμερα είναι η ελευθερία έκφρασης. Κοιτάξτε το καταστατικό. Λέει ελευθερία έκαρβασης. Αυτό είναι το βασικό. Θα ήθελα αυτό να σας το υπενθυμίσω όταν σκεφτούμε τις υποψηφιότητες και νομίζω υπάρχει μια σειρά υποψηφιότητων οι οποίες πραγματικά είναι άξιες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γιούρεκ, λέει Πρόεδρος. Δεν πρόκειται να σχολιάσω αρνητικά οποιαδήποτε υποψηφιότητα. Και αυτό γιατί η απονομή του βραβείου Ζαχάροφ αποτελεί μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να τιμηθούν αγώνες για τη δικαιοσύνη διαφόρων ειδών. Για να επανέλθω στα σχόλια του συναδέλφου, ωστόσο, να διευκρινίσω το εξή. Η Μέρι Βάγνερ έχει φορτωθεί ένα άδικο φορτίο πάνω της. Αποδέχεται τις άδικες κατηγορίες τις οποίες τις απαγγέλλονται, γιατί θεωρεί ότι είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να προασπίσει τις αρχές, τις αρχές που χαρακτηρίζουν τις χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη της Ρώμας και επίσης ε, σέβεται την αρχή του αλληλεοσεβασμού. Το δικαίωμα στη ζωή από τη σύλληψη είναι κάτι το οποίο κατοχυρώνεται και σταγματικά σε κάποιες χώρες. Η ζωή ξεκινά κατά την σύλληψη, πριν από τη γέννα. Και σε διάφορες περιπτώσεις ε, ακούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι, και η Ευρώπη είναι ουδέτερη στο θέμα αυτό. Δυστυχώ ο Καναδά όμω δεν είναι ουδέτερο. Καταπιέζεται την Μέρι Βάγνερ και νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει να τη δείξουμε αλληλεγγύη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Νομίζω ότι αυτό που χαρακτηρίζει μέχρι αυτή τη στιγμή τη διαχείριση του βραβείου Ζαχάροφ είναι πως είχαμε το σεβασμό από όλους προς όλες τις υποψηφιότητες και ήταν πάντα άτομα ακέραια, οργανώσεις σημαντικές που έχουν φημωθεί, καταπληκτικοί άνθρωποι που εργάζονται σε αδιανόητες συνθήκες για να σώσουν τους υπόλοιπους. Αλλά μπορεί να συμφωνεί κανείς γενικότερα ή όχι με τις υποψηφιότητε, συνήθως τις έχουμε σεβαστεί. Το πρόβλημα είναι ότι αν παρουσιάζεται μια υποψηφιότητα η οποία είναι μια άμεση επίθεση. Άμεση επίθεση. Μια απαράδεκτη χειραγώγηση, μια σχεδόν προσβολή για τις αξίες τις οποίες υπερασπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό πολλοί από εμά και κυρίως πολλές από εμάς να αισθανόμαστε ότι μας έχουν επιτεθεί και ότι διαμαρτυρόμαστε. Και αν συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε ένα κλίμα σεβασμού, γιατί το αξίζουν οι υποψηφιότητες, σας παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε πολιτικά και λαϊκιστικά κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό όσο το δικαίωμα της γυναίκας στην επιλογή. Κύριε Κούκαν. Δύο προτάσεις επιτρέψτε μου. Νομίζω ότι όλοι όλους μας απασχολεί το βραβείο Ζαχάροφ. Είναι δικαίωμα κάθε πολιτική ομάδας να υποβάλει τους υποψηφίου τους. Ζαχάροφ, ε, βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία έκφρασης. Είναι σημαντικό λοιπόν. Ενδεχομένω να υπάρχουν διαφορετικέ ερμηνείε για το τι σημαίνει ελευθερία σκέψη και έκφραση, αλλά όταν συζητάμε του υποψηφίου, θα προτιμούσα πραγματικά να υπογραμμίζεται η θετική πτυχή του κάθε υποψηφίου. Δεν ξέρω αν πραγματικά εδώ αρμόζει μια αρνητική καμπάνια. Ίσως θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε στα θετικά που θα σημάνουν και την νίκη στον διαγωνισμό αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βερζιά. Για την συνάδελφο Έλενα Βαλαντίνη να πω το εξή. Δεν είμαι βέβαιη ότι όλοι έχετε διαβάσει το καταστατικό του βραβείου Ζαχάροφ. Και διαβάστε το. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει τη το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία έκφρασης. Η ελευθερία του πνεύματος, όχι μόνο ελευθερία έκφρασης και σκέψης. Και ιδιαίτερως την πράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και κυρίως το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης. Αυτό μπορεί να είναι με τρόπο και αν υπάρχει πρόβλημα την προστασία των μειονοτήτων, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Νομίζω ότι κάποιες προτάσεις ε, είναι πραγματικά στο πνεύμα αυτό την σεβασμό του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας και νομίζω ότι και εδώ όλες οι υποψηφιότητες μπορούν να εξετάζονται. Όχι, δεν είναι μόνο η ελευθερία εκφράσης η οποία βραβεύεται με το βραβείο Ζαχάροφ, είναι μια έννοια πολύ πιο ευρεία. Και νομίζω ότι αυτό καλό θα ήταν να το υπενθυμίσουμε σε όλους τους συναδέλφους μας, να τους καλέσουμε να διαβάσουν το κανονισμό και το καταστατικό για το βραβείο Ζαχάροφ. Πρόεδρος, ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις. Και να δώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. It's time to uh, Σύντομα συμπεράσματα λοιπόν και αρκετές φορές κύριε Παντσέρη. Ξεκινώ με τις ευχαριστίες και εδώ ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έχουν υποβάλει υποψηφιότητες, όσους συμμετείχαν στη συζήτηση και επίσης όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι παρόντα ή που έχουν παρουσιάσει υποστήριξη κάποια υποψηφιότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Γερμηνείς. Δεν είναι μια συνηθισμένη συνεδρίαση αυτή και για μένα είναι η πρώτη φορά που είμαι συμπρόεδρος σε μια συνάντηση για το βραβείο Ζαχάροφ. Είναι πολύ ενδιαφέρον και επιτρέπει σε όλα τα μέλη να εξοικειωθούν με τις υποψηφιότητες και με το βραβείο το ίδιο. Για την ελευθερία της σκέψης, για την ελευθερία η οποία υπερβολικά συχνά πέφτει θύμα επιθέσεων σχεδόν παντού στον κόσμο τελευταία. Πριν να κλείσουμε τη συνεδρίαση, θέλω να σας υπενθυμίσω ποιο είναι το χρονοδιάγραφο. επέμενο βήμα για τη διαδικασία είναι η ψηφοφορία που θα έχουμε το σύντομο κατάλογο των τριών υποψηφιωτήτων. Θα γίνει την 3η 9 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες στην συνεδρίαση ΑΦΕΤ ΝΤΕΒΕ. Η διάσκεψη προέδρων θα αποφασίσει τον νικητή ή τους νικητές και θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα στις 25 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Ο νικητής θα προσκληθεί σε ανταλλαγή απόψεων σε μια κοινή συνάντηση που θα κάνουμε στις 20 στις 10 Δεκεμβρίου, με συγχωρείτε, ε, το Δεκέμβριο στο Στρασβούργο και η τελετή θα γίνει την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Στρασβούργο. Closed. Thank you again. Λύεται η συνεδρία. Σας ευχαριστώ.